να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην εξέλιξη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, μία αντίδραση στο ερώτημα της κυρίας Δεκάιζερ που μίλησε για την εκτέλεση του Βρετανού πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε ανεπιφύλακτα την εκτέλεση του Αχμαλσαϊ. Λυπούμεθα επίσης για το ότι η Κίνα δεν άκουσε τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενό κράτους μέλους για τη θανατική ποινή του Ιουσάη και για την αναβολή εκτέλεσής της. Ο πρώτος, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όμως ακόμα, ακόμα λέγω, απομείνει ένα σημείο στη μέση διάταξη. Παρακαλώ καθίστε. Καθίστε και κάντε ησυχία. Θα συζητήσουμε τώρα το ψήφισμα σχετικά με τις Φιλιππίνες. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια θλιβερή συνήθεια ε, αυτές ε, οι σειρές δολοφονιών με πολιτικά και θρησκευτικά κίνητρα. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, ναι. εντυπωσιαζόμαστε από τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκαν 57 ε, άτομα τα οποία είχαν διαπράξει το τρομερό αδίκημα του να υποβάλλουν και να στηρίζουν μία υποψηφιότητα Προέδρου. Πρόκειται για μία σφαγή εν ψυχρό από ένοπλες ομάδες ε, τις οποίες την έννοια δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Αυτή η δολοφονία η μαζική δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο σε αυτή τη χώρα η οποία γνωρίζει ε, δυστυχώς ε, ένοπλες εξεγέρσεις κυρίως στην περιοχή του Μιντανάου. Νομίζω ότι πέρα από, την, από τα συλληπιτήρια τα οποία θα πρέπει να εκφράσουμε για αυτά τα αιματερία γεγονότα, θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε μέσω συνεργασίας την ε, κυβέρνηση ε, των Φιλιππίνων να καταλάβουν με ποιο τρόπο μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει έτσι ώστε τέτοιου είδους ένοπλες αντιπαραθέσεις να σταματήσουν να αιματοκυλούν αυτήν τη δύστιχη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέστλερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, η σφαγή στις 23 Νοεμβρίου πέρσι στην Μεγκαντινάου στις Φιλιππίνες ήταν μαύρη μέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια άνω των 70 νεκρών και ως ε, δημοσιογράφος μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως 30 από αυτούς νεκρούς ήταν δημοσιογράφοι σύμφωνα με το International Crisis Group δεν έχουν δολοφονηθεί ποτέ τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι με ένα χτύπημα. Θεωρούμε λοιπόν πως θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται αυτό στο σημερινό μας ψήφισμα. Επίσης, εμείς θέλουμε ως ΕΛΚ να γίνει πιο έντονο το ψήφισμα και έχουμε ζητήσει χωριστή σφοφορία σε τρία σημεία. Γι' αυτό ζητάμε εκ μέρους ε, του ΕΛΚ ειδικά να καταψηφιστεί το εκτιμώντας F καθώς καταγγέλει τις ε, Φιλιππίνες και στο σημείο 2 εκεί πέρα που αναφέρονται οι υποτιθέμενες καθυστερήσεις έρευνες επίσης να φύγουν επίσης και για τους εξαφανιστέντες σε ε, φιλιππινέζικες φυλακές και αυτό δεν έχει ε, τεκμηριωθεί ως κατηγορία και πρέπει να διαγραφεί. Ένα λεπτό κύριο Στάνο, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το έγκλημα του Μιντανά θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφαστα διότι αποδεικνύει το πόσο σε ορισμένα ε, μέρη των, των Φιλιππίνων δεν υπάρχει νόμος και τάξη. Ε, δεν υπάρχει σειρή κυβέρνηση, υπάρχει διαφθορά και φτώχεια. Ε, γι' αυτό και όλα αυτά ενθαρρύνουν την Αλκάιντα στο νότιο μέρο του νησιού. Έχει πολιτικά κινήτρα αυτό το έγκλημα, οπότε θα πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και το ιστορικό πλαίσιο δεν θα πρέπει βέβαια να υποτιμούμε τι προσπάθειε τη κυβέρνηση, ώστε να ε, υπάρχει επιτέλου δημοκρατία μετά από 25 χρόνια κατόπιν τη πτώση τη δικτατορία του Μάρκο. Ούτε να υποτιμούμε την απειλή της τρομοκρατίας της ομάδας Σαγεύ. Υπάρχει δημιουργική προσπάθεια. Θα πρέπει να παρασχεθεί αρρωγή στη χώρα αυτή. Γιατί έχουμε κοινέ αξίε με αυτή τη χώρα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε να αποκτήσει το κράτο δικαίου σε κεντρική, σε κυβέρνηση, αλλά και αυτοδιοίκηση. Ο κύριο Ταραβέλ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τον προηγούμενο Νοέμβρη είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την ε, κυρία Ερίτα Μπούργος, την ε, μητέρα του νεαρού Μπούργος, ο οποίος απήχθη ε, στις 28 Απριλίου του 2007 από μια ένοπλη ομάδα σε ένα πολυσύχνωστο εμπορικό κέντρο της Μανίλας και έκτοτε αγνοούνται, αγνοείται η τύχη του. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι εξαφανισμένοι απαχθέντες Φιλιππινέζοι Ε, εν ώψη των εκλογών του Μαΐου 2010 φοβούμεθα αναζωπήρωση το, το, της ε, τάσης αυτής και επομένως θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Επίσης ε, καταδικάζομαι την ένοπλη επίθεση και την σφαγή στην περιοχή Μαγκίντα καθώς επίσης και για τον βασανισμό του Ισμαήλ Μαγκούντα Νάο. Ευχαριστούμε κύριε Και τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλο ο κόσμος ελπίζε ε, να έχουμε δημοκρατικές εξελίξεις ε, στις Φιλιππίνες και αυτό μέχρι από μία εικοσαετία περίπου. Τώρα έχουμε τώρα τα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ελπίδες για καλύτερη τύχη και των εργαζόμενων και όλο το λαό γενικότερα. Υπήρχε μια δημοκρατική ομαλότηση, υπήρχαν ε, νόμιμες εκλογές, όμως μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί ανισχυτικά μηνύματα όσον αφορά τη διαφθορά, τη βία, ε, τις νόθες εκλογές Και εκδήλωση αυτών των φαινομένων είναι αυτό το πήγαινε στο Μιντανά. Όλες αυτές οι πράξεις κατά της αντιπολίτευσης που έχουν γίνει αυτή η επίθεση της ένοπλης ομάδας που δράσει στην περιοχή αυτή. Είχαμε 30 ανθρωποκτονίες στην περιοχή ε, έγινε σφαγή μπορούμε να πούμε δημοσιογράφων κάτι το οποίο αποτελεί ρεκόρ δεν θα πρέπει κάτι τέτοιο να το παραβλέψουμε δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πειραθεί η κατάσταση στη φίλη Φιλιππίνες θα πρέπει να ξαναγίνει η χώρα παράδειγμα προς μίμηση όπως ήταν ε, μέχρι πριν από μια εικοσαετία Θα πρέπει να δείξουμε ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τι εξελίξει στη χώρα. Για ένα μισό λεπτό, λέει Ο πρόεδρο έχει το λόγο η κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφορμή του ψηφίσματός μας απετέλεσε η παραβαρή δολοφονία 77 ανθρώπων που πήγαν να εγγραφούν για να υποστηρίξουν μία υποψηφιότητα και βεβαίως ήταν εκεί παρόντες και της, ε, άτομα και της τοπικής αστυνομίας. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των εξοδικαστικών εκτελέσεων με πολιτικά κέντρα, κίνητρα τα οποία ποτέ δεν εξηχνιάζονται. Η κυβέρνηση δεν έδειξε καμία θέληση να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Σε εκατοντάδες περιπτώσεις είχαμε τέτοιες ολοφονίες, δύο μόνο εξεχνιάστηκαν, κανένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος δεν τιμωρήθηκε. Ο δε ειδικό αποσαλμένος του ΟΗΕ λέει πως ε, έχουν εξαφανιστεί μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή συνδικαλιστές και όσοι είναι υπέρ του αναδασμού. Έχουν τρομάξει τις ε, εκπροσώπους ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών και περιορίζουν την πολιτική δραστηριότητα στην χώρα και φοβόμαστε πως θα οδηγηθούμε και σε περισσότερες πολιτικές δολοφονίες. Γι' αυτό είναι απολύτως κατεπήγον η κυβέρνηση των Φιλιππινών να αναλάβει μέτρα αποτελεσματικά και θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6 λέει να απελευθερώσει όσοι είναι ακόμα κρατούμενοι θέλουμε αυτό να αντικατασταθεί με το να καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίσει όλοι όσοι έχουν απαχθεί να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Λοχμπίλερ και τώρα οι ομιλητέ των πολιτικών ομάδων ξεκινούμε με του σοσιαλιστέ δημοκράτε. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Παλέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν ρωτήσετε το μέσο Ευρωπαίο για το τι συμβαίνει στις Φιλιππίνες, δεν θα λάβετε και καμία απάντηση. Δεν τα δείχνει η τηλεόραση, είναι ήσυχα τα πράγματα άρα, αλλά οι πολιτικές αυτές φαγές ε, ταφές ζωντανών ανθρώπων ε, εκτελέσει με φρικιαστικούς τρόπους είναι καθημερινή κατάσταση τώρα δολοφονήθηκαν 77 άτομα η μισή από τους οποίους ήταν ε, δημοσιογράφοι και μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιογράφων που εκτελέστηκε με μιας Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση να σταματήσει αυτά τα φρικτά εγκλήματα θα πρέπει να διαλύσει αυτές τις παραστρατιωτικές ομάδες και να θέσει τέλος στην ατιμορρησία εν και των εκλογών που έρχονται. Ευχαριστώ. Κύριε και σε ευχαριστούμε. Και τώρα οι υπόλοιποι αγορητές. Για ένα λεπτό έχει το λόγο κυρία Γκέριγκερ Ντε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 10 Μαΐου έχουμε προεδρικές αλλά και δημοτικές εκλογές. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε οι εκλογές αυτές να είναι δίκαιες. Θα πρέπει μένω σε περίβαση να καταδικάσουμε τους ε, ένοχους της εν λόγω σφαγής. Μέχρι σήμερα πάντως η δικαιοσύνη κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα λάθη όσον αφορά τις σχετικές έρευνες. Επομένως η παρανομία θα συνεχίσει να βασιλεύει στη χώρα. Θα πρέπει οι Φιλιππίνες να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί αυτά τα χρήματα δόθηκαν ούτως ώστε να οικοδομηθεί κράτος δικαίου και δημοκρατία στη χώρα. Ευχαριστούμε Και τώρα, κάτσε μόνο δύο συναδελφούς το λόγο και για ένα λεπτό έχει ο κύριος Ρωμέρα το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομα. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τώρα ε, έχει έρθει μια καινούργια χρονιά, έχουμε μια καινούργια συνθήκη. Όμως, όμως οι κακές συνήθειες ε, παραμένουν ε, γιατί συνεχίζει να απουσιάζει το Συμβούλιο σε τέτοιου κατεπίγουσε κατεπίγουσες συζητήσεις. Επίσης ε, δεν υπάρχει ούτε ένας διοργανικός διάλογος τόσο να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση των Φιλιππίνων, σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι παρά την κατάσταση αυτή και την ΑΕΤ έχουμε πάνω από χίλιου νεκρού κάθε χρόνο. Επομένω το πρόβλημα είναι δομικό εδώ πέρα και άρα χρειάζεται δομικά διαρθωτικά μέτρα. Δεν είναι δυνατόν πάντοτε να μα κινητοποιούν τα πρωτοσέλιδα. Βλέπουμε ότι αυτοί που χτυπιούνται πρώτοι είναι δημοσιογράφοι, είναι αυτοί που έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα δεν μπορούμε να, να ε, σιωπούμε, θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί μπροστά σε τέτοιε κρίσει. Ευχαριστούμε κύριε Ρομέρα, λέει και τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Τσαρνέτσκι. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όμως το Συμβούλιο και συγκεκριμένα η Ισπανική Προεδρία δεν αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρονται για ανθρώπινα δικαιώματα γιατί απουσιάζουν από την αίθουσα μια που συζητούμε τέτοια ζητήματα. Εμείς θα συζητούμε αλλά αυτοί δεν ήρθαν στη συζήτηση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Οι Φιλιππίνες είναι χώρα χριστιανική, χριστιανική παράδοση. Συμμερίζονται μαζί μας αξίες ευρωπαϊκές. Άρα θα πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται. Θα πρέπει επομένω ξεκάθαρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς εκείνους οι οποίοι υποφέρουν στη χώρα εκείνη. Αυτή είναι καθήκον μας. Ο πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα εσείς το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ την ύπατη εκπρόσωπο και κατ' επέκταση βεβαίως και την Επιτροπή. Η ε, σφαγή ε, στο Μαγκίντα Ναό στις 23 Νοεμβρίου του 2009 ε, κατά τη διάρκεια του οποίου δολοφονήθηκαν βάναυσα 57 ε, μέλη ε, της αυτοκινητοπομπής βεβαίως αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες και προστίθενται στις απαγωγές, εκτοπισμούς, εξοδικαστικές διαδικασίες στην χώρα αυτή. Βεβαίω ελήφθησαν άμεσα μέτρα ε, έτσι ώστε να προσαχθούν ενώπιον τη δικαιοσύνης ε, ε, οι υπεύθυνοι και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η γνώση της ατιμορρησίας στην χώρα αυτή. Κύριε Πρόεδρε, ελήφθησαν από πλευρά τη κυβερνήσεω κάποια σημαντικά μέτρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα η πρόεδρος ε, Αρόγιο ε, ακύρωσε την ε, θανατική πίνη και προσυπέγραψε την Ασιατική Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης ελπίζομαι ότι ε, βάσει μιας ε, συμφωνίας ειρήνης ε, που θα είναι εποφελής και προς τα δύο μέλη θα ολοκληρωθεί μια τεσσαρακονταετής ένοπλη σύραξη στην περιοχή του Μαγκιντανάου θρησκευτικού χαρακτήρα. Πιστεύομαι ότι η περίπτωση του Μαγκίντα πρόκειται στην ουσία για ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών φατριών και συγκεκριμένα πολιτικών οικογενειών και επομένως δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, πολιτικών αντιπαραθέσεων. Διαπραγματευόμαστε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην, και την κατάστασή τους στις Φιλιππίνες. Επίσης, διαπραγματευόμαστε συμφωνία χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στήριξης της δικαιοσύνης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, σε συμφωνία με την ε, κυβέρνηση, έχουμε ε, ξεκινήσει ε, μια αποστολή όσον αφορά την στήριξη της δικαιοσύνης στις Φιλιππίνες. Και αυτό, αυτή η αποστολή περιλαμβάνει στήριξη έργου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Ομάδων Κοινωνίας των Πολιτών και επίσης θα είναι επιφορτισμένο παρακολούθηση της πρόοδου της χώρας όσον αφορά την καταπολέμηση εξοδικαστικών εκτελέσεων και E Το EPJUST ε, θα έχει μια αρχική διάρκεια 18 μηνών ε, και ε, θα μπορεί να επιμηκυνθεί βάσει των αποτελεσμάτων του. Επίσης, έχουμε και άλλα υφιστάμενα προγράμματα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία προσπαθούν να ενισχύσουν τη θέση, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή δεσμεύσεις, ε, πράξεις ε, στήριξης ε, της υπογραφής διεθνών συνθήκων. Επίσης, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στην διαδικασία ειρήνευσης ε, της ε, περιοχής Μαγκίντα βάσει της νέας συμφωνίας και βάσει των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όμως κύριε Πρόεδρε είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ακόμα περισσότερο όσον αφορά την χώρα αυτή εάν οι μέχρι τώρα διαδικασίες στεφθούν από επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Υπενθυμίζω στην κυρία Λοχβίλερ ότι θα πρέπει να μην ξεχάσει να υποβάλει την κατάλληλη στιγμή της διαδικασίας την προφορική της τροπολογία.